Ναι, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της Ιζαμπέλ Τομάς σχετικά με το πώς θα καταστούν ομοιόμορφοι έλεγχοι της αλίας στην Ευρώπη. Δίνω τον λόγο ε, στην κυρία Τόμας ε, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε.